να αποφαθεί και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσο γίνεται. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρία, λέει ο Πρόεδρο. Ε, αύριο το πρωί, επόμενη συνεδρίαση από τι 9 μέχρι τη 1 και το απόγευμα από τι 3 μέχρι τι 10 το βράδυ. Θα βρείτε την ημερήσια διάταξη και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Λίγη τη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ πολύ.